να διασφαλίσει ότι αυτοί οι οποίοι υπεξαίρεσαν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία δεν θα μείνουν ατιμόρυτοι. Ευχαριστούμε. Κύριε Επίτροπε, υπάρχουν έξι ψηφίσματα. Η συζήτηση έληξε και θα ψηφίσουμε αύριο στις 12 το μεσημέρι. Τώρα, Τώρα η μερίσια διάταξη προβλέπει την έκθεση πρόοδο 2012 για την Βοσνία και Ερζεγοβίνη. Το λόγο έχει η Υπουργό Κρήτον. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι προβουλευτέ, οι εξελίξει στη Βοσνία και Ζεγοβίνη δεν έχουν ακολουθήσει το ρυθμό που ελπίζαμε και προσδοκούσαμε. Υπάρχουν διάφορε ανησυχίε και ξέρω ότι τι συμμερίζεται και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έτσι όπω φαίνεται και από την πρόταση ψηφίσματο που θα ψηφίσετε αύριο. Επιτρέψτε μου να υποφελθώ από την ευκαιρία αυτή για να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα την Doris Πακ για την δέσμευση που έχει αναλάβει, για τις γνώσεις της επίσης που τις χρησιμοποίησε ως εισηγητής σας. Ιδιαίτερα θέλω εδώ να τονίσω την θετική επιρροή που μπορείτε να έχετε στις εξελίξεις στη Βοσνία Ζεγοβίνη. Το Δεκέμβρη μας πέρασε το Συμβούλιο σημείωσε κάποια πρόοδο στη Βοσνία Ζεγοβίνη ήδη επειδή το αρχές του 2012 φτιάχτηκε το πρώτο σε επίπεδο κράτου Συμβούλιο Υπουργών. Επίσης, ε, εκφράσαμε την ικανοποίησή μας από την έγκριση δύο νόμων ε, εκείνων για τις κρατικές ενισχύσεις και εκείνων για την υπογραφή. Δυστυχώς όμως ο ρυθμός δεν κρατήθηκε όπως τον περιμέναμε και έτσι έγιναν καθυστερήσεις. Και απογοητευτήκαμε επίσης από την πρόοδο που επιτεύθηκε όσον αφορά ε, τα θέματα που είχαμε στην ατζέντα. Και επειδή εξακολουθούσε να υπάρχει διχαστική ρητορική στη χώρα. Το Δεκέμβριο επίση το Συμβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του επειδή ξεκίνησε ο διάλογο υψηλού επίπεδου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την διαδικασία ένταξη τη Βοσνία Ερζεγοβίνη με εκπροσώπου πολιτικού από τη χώρα αυτή. Μία από τι προτεραιότητε πάντω για τη Βοσνία Ερζεγοβίνη είναι να συμμορφωθεί το Σύνταγμά τη με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την δικαστική απόφαση Φέτζικ Φίντσι πρέπει να δούμε αποδείξεις για αλλαγές προς την κατεύθυνση αυτή που θέλουμε. Πρέπει να εφαρμοστεί η συμφωνία Σέτσικ Φίντσι, η απόφαση αυτή δηλαδή. Επίσης, η Βοσνία πρέπει να αποδείξει ότι ικανοποιητικά ακολουθεί την πορεία εφαρμογών των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει σύμφωνα με την Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. Αυτά είναι στοιχεία κλειδί που πρέπει ρεαλιστικά να προχωρήσουν προκειμένου να συζητήσουμε την ε, προσχώρηση της χώρας αυτής. Το Συμβούλιο επίσης έχει υπογραμμίσει τη σημασία που έχει να υπάρξει αποτελεσματικός συντονισμός των ε, υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η χώρα απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς έχουμε επαναλάβει την στήριξή μας στο διαρθρωμένο διάλογο για την δικαιοσύνη στα πλαίσια της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και έχουμε ζητήσει από όλες τις αρχές της Βοσνίας Ζεγοβίνη να συμμετάσχουν υποκοθομητικά στη διαδικασία αυτή. Το στοιχείο κλειδί για να διασφαλίσουμε την παγίωση ενός ε, ανεξάρτητου, αμερόληπτου και αξιόπιστου δικαστικού συστήματος. Πρόεδρε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ, η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να συνεχίσει να ενισχύει τη στήριξή τη στην διαδικασία ολοκλήρωση τη Βοσνία και Ζεγοβίνη. Είναι μέρο μια διαδικασία που έχει επιβεβαιωθεί και έχουμε βεβαιώσει και την απόλυτη στήριξή μα. Όμω η πολιτική ηγεσία στη Βοσνία Ζεγοβίνη πρέπει να διδικοποιήσει τι προσπάθειε. Οι υποχρώσει που έχουν αναλυφθεί πρέπει να καλυφθούν και επιπλέον δουλειά απαιτείται για να υπάρξει μεγαλύτερη σταθερότητα και ευημερία στην χώρα η ηγεσία το φίλει αυτό στους πολίτες της που αξίζουν ένα καλύτερο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο Επίτροπος Φίλου έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, Υπουργοί. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, κυρία Ντόρι Σπακ ε, πρώτα απ' όλα. Είναι εξαιρετική η έκθεση που συνέταξε για τη Βοσνία Ζεγοβίνη. Πέρυσι σας είπα ότι όταν μιλάμε για την βοσνια ζεγοβινη είναι δύσκολο να κάνουμε μια συνολικά θετική αποτίμηση. Δυστυχώς το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζω και φέτος. Όπως βλέπουμε στο σχέδιο έκθεσης και πάλι είναι μάλλον περιορισμένη η πρόοδος δεν υπάρχει ε, ένα γενικότερο όραμα για τον προσανατολισμό που ακολουθεί η χώρα. Ε, όπως βλέπουμε και στο ψήφισμα, η χώρα ε, παραμένει ουραγός σε σχέση με άλλες γειτονικές ε, χώρες. Ε, έχει βέβαια ενταθεί η δέσμευσή μας ε, για την Βοσνία Ζεγοβίνη και έχουν ενταθεί και πολιτικές προσπάθειες σε όλα τα επίπεδα τους ε, τελευταίους μήνες. Κλιμακώθηκε η διπλωματική δραστηριότητα στην περιοχή για να λυθούν τα πλέον επίγοντα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα. Για να μην πολυλογώ, ε, για να εφαρμοστούν όλα τα μέτρα στον οδικό χάρτη που συμφωνήθηκαν ε, τον Ιούνιο του 2012 από ε, τις πολιτικές αρχές και αναφέρονται επίσης στην έκθεσή σας, στο ψήφισμά σας μάλλον και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Αυτό θα πρέπει να κάνουμε, να συζητήσουμε το θέμα της υπόθεσης του διότι εάν μέσα από τη διαδικασία διευκόλυνσης παρόλα αυτά δεν έχουμε αυτά αποτελέσματα, θα πρέπει να ακυρωθεί ο τρίτος γύρος του διαλόγου υψηλού επίπεδου για την διαδικασία σύνδεσης. Θεωρούμε ότι κάποιοι πολιτικοί ενδιαφέρονται περισσότερο για εθνοτικά συμφέροντα παρά για την απόφαση Σέντιτς Φίνσης. Η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μόνο μπορεί να βοηθήσει. Η πολιτική ηγεσία του τόπου είναι εκείνη που μπορεί να ε, αναλάβει πραγματική δέσμευση. Η πολιτική αστάθεια στην Ομοσπονδία που επικρατεί σήμερα καθιστά δύσκολη την εξέβρεση μια συμβαστική λύση για τόσο δύσκολα ζητήματα. Παρόλα αυτά είναι ζωτική σημασία στο να συμβεί αυτό. θα γίνει Μεσα γειτονική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, η Βοσνία Ζεγοβίνη να προχωρήσει τη διαδικασία. Ελπίζουμε να ε, στεφθεί με επιτυχή η διαδικασία και για τα δύο μέρη με τους πρώην ε, πρωθυπουργούς Βοσνίας Βοσνίας-Ζεγοβίνης και της Κροατίας. Συσκέφθηκα δύο φορές για αυτό το θέμα. Επίσης είχαμε πέντε τεχνικές συσκέψεις υπηρεσιακές ε, και παρά τις επαναλαμβανόμενες αποτυχίες εμείς ε, τονίζουμε ότι η πάγια δέσμευσή μας και η υποστήριξή μας είναι στη διάθεση ε, όλων όσων επιτόπου επιθυμούν να σημειωθεί η πρόοδος στο δικαστικό σύστημα. Έχει αποφέρει καρπούς η προσπάθειά μας και πιστεύω ότι ένθερμα όλοι υποστηρίζουμε τη διαδικασία όπως και εσείς κυρία Πάκη θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ευχαριστήσω όλους ιδιαίτερες κλειώδες στην παρέμβαση μου. ευχαριστώ μου από πλευρά των πολιτικών ομάδων ακούμε στους μεμονωμένους ομιλητές η κυρία Πάκα από πλευρά του ΑΛΚ δύο λεπτά Ευχαριστώ Κυρία Πρόεδρε κύριε φίλε Και τέσσερι εβδομάδε έχουμε αναβάλει αυτήν την συζήτηση, Ελπίζοντα ότι κάτι θετικό θα συμβεί σε αυτή τη χώρα. Δυστυχώ όμω δεν συνέβη, τίποτα δεν βελτιώθηκε δεν υπάρχει συμφωνία, δεν υπάρχει καμία κυβέρνηση που να μπορεί να δράσει και ο πρόεδρος σήμερα βρίσκεται σε μια κατάσταση παραλυσίας θα έλεγα χωρίς να του επιτρέπεται να δραστηριοποιηθεί. Επίσης όσον αφορά την αντιπολίτευση πάλι μπορούμε να πούμε ότι τίποτα δεν γίνεται. Η κατάσταση είναι πραγματικά απογοητευτική στη Βοσνία Ζεγοβίνη. Η πολιτική εκτός της ε, Βοσνίας Ζεγοβίνης η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθούν να βοηθήσουν να βελτιωθούν τα πράγματα. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι υπάρχουν όμως σημάδια που μας κάνουν πραγματικά να ανησυχήσουμε εξαιρετικά. Θεωρώ πραγματικά ότι είμαστε υποχρεωμένοι να στηρίξουμε τους πολίτες αυτής της περιοχής και να τους δώσουμε δυνατότητες να εποφεληθούν και να μην είναι θύματα αυτής της απραξίας και ανικανότητας που επικρατεί. Θα ήθελα πραγματικά να πω ότι ο λόγος για τον οποίο έφτασα σε αυτά τα συμπεράσματα είναι ότι σήμερα δεν υπάρχει ούτε ένας πολίτης που να αναγνωρίζει την θετική δράση των πολιτικών. Θα πρέπει βέβαια εμείς να πούμε την αλήθεια στους ε, πολίτες των χωρών μας. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να μεταφέρουμε κονδύλια στην περιοχή αυτή, ενώ διαρκώς συνεχίζουν να μας κοροϊδεύουν οι, πολίτες, οι πολιτικοί συγγνώμη, της χώρας αυτής. Νιώθω πραγματικά ότι εδώ και 23 χρόνια έχουμε δεσμευθεί προς τους πολίτες της Βοσνίας της Και αν υπήρχε καλή διακυβέρνηση θα είχαν μια εργασία, οι πολίτες αυτής της χώρας και τα παιδιά θα μπορούσαν να πάνε σε ένα σχολείο και να μορφωθούν. Πιστεύω ότι πραγματικά οφείλουμε αυτούς τους πολίτες της Βορδίας Ζεγοβίνης. Ευχαριστώ πολύ. Η... η κυρία Μπόσκουρτ. Έχουν περάσει οι προθεσμίες, προσπάθειες γίνονται, παρόλα αυτά χωρίς αποτέλεσμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε να πούμε ποτέ ότι είναι σωστές οι εκλογές εφόσον δεν υπάρχει ελεύθερη αντιπροσώπευση. Είναι πολύ βασικό. Γι' αυτό και η απόφαση Σέντιτς Φίντσι είναι καθοριστική. Είμαι και εγώ από τους άλλους. Θυμάμαι ότι είχατε πει μια, είχε πει ότι μια φορά θα μπορούσε να είναι πρόεδρος της χώρας. Εγώ δεν μπορώ να στηρίξω πάντως ε, την ε, πρόταση που λέει ότι πρέπει να ε, υπάρξει διακοπή της συμμετοχής στο Συμβούλιο της Ευρώπης της Βοσνίας της Ζεγοβίνης. Μπορεί να μην συμμετέχει, αλλά τι θα γίνει με τις άλλες χώρες. Οι συνέπειες θα είναι μεγάλες για τη Βοσνία ριζεγοβινη Κροατία και Βοσνία ριζεγοβινη πρέπει να βρουν τρόπους να τα βρουν, όχι να χωρίσουν ακόμα περισσότερο. Οι πολίτες της Βοσνίας Ερζεγοβίνης είναι αυτοί οι οποίοι υποφέρουν από την ανεργία και από την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Οι περισσότεροι θέλουν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλουν την προστασία της. Η τάση αυτή μειώνεται. Είμαστε σε διέξοδο. Δεν αλλάζουν τα πράγματα στη Βοσνία, ούτε και η Κομισιόν ε, αλλάζει τίποτα. Στην περιοχή όμως τα πράγματα αλλάζουν. Η Κροατία εμποδίζει τους πολίτες να ταξιδεύουν της Βοσνίας Ριζεγοβίνη, την αυτοτιμωρία στη Βοσνία ριζεγοβινη και ισχύει. Ερώτηση είναι αυτή. Έχουμε την ευθύνη για τα Δυτικά Βαλκάνια. Οι εξελίξεις στη Βοσνία Ζεγοβίνη επηρεάζουν ολόκληρη την περιοχή. Πώς θα διασφαλίσουμε λοιπόν βιωσιμότητα και σταθερότητα στην περιοχή. Αν υπάρχει θέληση σίγουρα θα βρεθεί και ο τρόπος. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε εκ μέρους των φιλελεύθερων η κυρία Νέιτς Άιτονμπρουκ. Δύο λεπτά παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Προεδρεύουσα του Συμβουλίου, κύριε Πίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, Αντιλαμβάνομαι την απελπισία σας που τόσα πολλά χρόνια βλέπετε τις εξελίξεις στη Βοσνία Ρισεχοβίνη να μην φέρνουν αποτελέσματα παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει για να βελτιωθεί η κατάσταση εκεί. Και τώρα για άλλη μια φορά βλέπουμε ότι δεν τηρούνται οι προθεσμίες. Αντιλαμβάνομαι την κυρία Πακ η οποία έχει πολύ ταπεραμέντο, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι πολύ δυναμική. Καταλαβαίνω λοιπόν από την απελπισία αυτή προτείνει τροπολογία με την οποία ζητάει να, από το, να αποκλειστεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης, να αποβληθεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης η χώρα. Μπορώ να τα καταλάβω όλα αυτά, αλλά δεν συμφωνώ. Και δεν συμφωνώ γιατί όσο περισσότερες δυσκολίες παρουσιάζει η Βοσνία Αρζεγοβίνη, τόσο περισσότερα μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης θα ζητήσουν την, τον αποκλεισμό αυτό. Παρ' όλα αυτά αυτό θα χειροτερέψει ακόμα περισσότερο την κατάσταση της χώρας. Γι' αυτό και δεν συμφωνώ με την αποβολή. Αντίθετα, πιστεύω ότι πρέπει αντί να βάζουμε μεγάλους όρους, να βάζουμε μικρούς. Ο Λαφοντέν ε, τα έχει περιγράψει αυτά στους διάφορους μύθους του. Πρέπει να επιμείνουμε απέναντι στη Βοσνία Ζεγοβίνη και η τροπολογία της κυρίας Πακ πιστεύω ότι δεν έχει θέση εδώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τους πράσινους. Η κυρία Κορνέλησεν για 1,5 λεπτό. Πρόεδρε. Yeah, I have a mic now. Uh, since it... Συγγνώμη που είσαι διακοπή μικροφώνου. Από χτες έχουμε ξεκινήσει τη συζήτηση εάν η χώρα αυτή. Η κυρία Πακ προτείνει να ζητήσουμε από το Συμβούλιο της βοσνιας ερζεγοβινης καθοτι δεν εχουν τηρησει καμια μα καμια προθεσμια οσον αφορα τις συνταγματικέ μεταρρυθμισεις που χρειαζεται επιγοντως η χωρα αυτη η κυρια πακ προτεινει να αποκλείσει προσωρινά την Βοσνία Αρζεγοβίνη από την συμμετοχή της σε αυτό και δεν πιστεύω ότι πρέπει να διακόψουμε τουλάχιστον την δική μας χρηματοδότηση. Γι' αυτό και πιστεύω τα δύο θέματα πρέπει να αποφασιστούν ξεχωριστά. Θα ζητήσω λοιπόν ξεχωριστή ψηφοφορία. Υπάρχει βεβαίως ε, εδώ η ανάγκη οι πολιτικοί ηγέτες της Βοσνίας Ερζεγοβίνης να απαντήσουν για την εγκληματική τους απραξία. Επίσης είναι επίγον η διεθνής κοινότητα να δράσει και αν τελικά απαγορευτεί η συμμετοχή της ε, Βοσνίας Ερζεγοβίνης, καμία χώρα πλέον δεν πρόκειται να λάβει τα μέτρα αυτά τα οποία πρέπει να λάβει αν υπάρχουν τέτοιες επιπτώσεις. Βεβαίως και πρέπει να αλλάξει η κατάσταση στην Βοσνία Ζεγοβίνη και εμείς θα πρέπει ενδεχομένως να σταματήσουμε να εθελοτυφλούμε και να κοιτάξουμε τις πραγματικές ανάγκες και πώς μπορούμε να στηρίξουμε τους πολίτες της Βοσνίας της Μπορείτε να απαντήσετε ερώτηση, υπάρχει μπλε κάρτα. Μάλιστα. Κύριε Κονέλισεν, ακούγοντας αυτά που μόλις είπατε, Ερωτώ, πώς δικαιολογείται τα ουσιαστικά ποσά, κονδύλια που έχουν σταλεί στην Βοσνία Ζεγοβίνη μάλλον από την Βοσνία Ζεγοβίνη στην εκλογική σας ε, περιφέρεια. Κοιτάξτε, η Βοσνία Ζεγοβίνη, οι πολίτες της Βοσνίας Ζεγοβίνης είναι Ευρωπαίοι πολίτες και θα έπρεπε να ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόοδος που έχει επιτευχθεί εκεί είναι και δική μας πρόοδος. Όλα τα χρήματα λοιπόν που δαπανώνται για την ανάπτυξή τους, για τις υποδομές τους και για κοινωνικά θέματα όπως η απασχόληση, για την καταπολέμηση της ε, φτώχειας, ουσιαστικά θα είναι προς όφελος όλων των πολιτών της Ευρώπης. Δεν πρόκειται για φιλανθρωπία, πρόκειται για αλληλεγγύη. Σας ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Πορεύα. από τους Ευρωπαίους Συντηρητικούς. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, για άλλη μια φορά εξετάζουμε τον τρόπο με τον οποίο προχωράει η Βοσνία Ζεγοβίνη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πρέπει να πω ότι είναι ο πιο δύναμος κρίκος των Δυτικών Βαλκανίων. Οι αρχές της χώρας πρέπει να επικεντρωθούν πολύ σοβαρά στην καλή διακυβέρνηση, στο κράτος δικαίου, στην οικοδόμηση δημοκρατικών θεσμών, στην δημιουργία ενός ανεξάρτητου δικαστικού συστήματος, και να προχωρήσουν σε οικονομικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις, αλλά να καταπολεμήσουν και την ανεργία. Υπάρχει και το πρόβλημα της διαφθοράς, το οποίο είναι παρόν παντού στη δημόσια ζωή της χώρας. Όπως επίσης υπάρχει και το θέμα της εμπορίας ανθρώπων. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει πλουραλισμό στα μέσα ενημέρωσης επίσης και υπάρχουν και εθνικές διαμάχες, εθνοτικές. Νομίζω λοιπόν ότι η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ θα ήταν μια πολύ μεγάλη επένδυση. Συνεπώς η Βοσνία Ερσεγοβίνη θα έπρεπε να τηρήσει τα κριτήριά μας. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Μπέλντερ. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Στις 7 Μαΐου πήρα από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μια καθισχαστική απάντηση στην ερώτησή μου που ρωτούσαν οι δραστηριότητες ε, του Ιράν και των Βαχαμπιστών ε, λαμβάνουν χώρα στην Βοσνία Ερζεγοβίνη. Και μια εβδομάδα αργότερα η βοσνική κυβέρνηση έδιωξε δύο εξέχοντες ε, πρέσβεις από το Ιράν που βρίσκονταν στο Σαράγεβο ε, λέγοντας ότι πρόκειται για κατασκόπους. Και μάλιστα υπήρξαν και φωτογραφίες στον τύπο που έδειχναν τους δύο αυτούς διπλωμάτες πώς έφευγαν εφόσον είχαν αποκαλυφθεί ότι ήταν κατάσκοποι. Περιμένω λοιπόν μια σοβαρή απάντηση αυτή τη φορά. Θα προσπαθήσω και πάλι, κάνω μια δεύτερη απόπειρα. Λοιπόν, πιστεύετε ότι η διαδικασία ολοκλήρωσης στην Βοσνία συνάδει, είναι συμβατή με τις στενές επαφές και τη συνεργασία που έχει ο πολιτικός κόσμος με το θρησκευτικό establishment στο Σαράγεβο και τους Ισλαμιστές από το Ιράν. Επίσης πιστεύετε ότι η παρουσία βαχαμπιστών στην Βοσνία ε, αποτελεί ή όχι κίνδυνο για την χώρα και την περιοχή ολόκληρη τη στιγμή που δραστηριοποιούνται εκεί παρά τους νόμους της χώρας. Ο κύριος Αγκουράκης τώρα έχει το λόγο εκ μέρους της ΓΟΕ. Ένα λεπτό. Μετά την ένταξη ακόμα μιας ταλαιπωρημένης χώρας στην κόλαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα εντείνει την εκμετάλλευση των εργαζομένων για να διασφαλίσει την κερδοφορία των μονοπωλίων, τα γεωστρατηγικά και ενεργειακά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ζητάει επίσης επιτάχυνση των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων για να θεραπευτούν δήθεν οι πολλές πληγές που δημιούργησε ο πόλεμος του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Αμερικανών ενάντια στο Ιουγκοσλάβικο λαό και η υπεριαλιστική ειρήνη που ακολούθησε συνιστά πρόκληση να απευθύνουν συστάσεις για τις εθνοτικές διαιρέσεις τη διαφθορά την ανεργία την απίστευτη φτώχεια τους χιλιάδες πρόσφυγες αυτοί που τα δημιούργησαν η ευρωπαϊκή ένωση και το πολιτικό της προσωπικό. πάει πολύ να εμφανίζεται τιμητής η ευρωπαϊκή ένωση που διαμέλυσε τη γιουγκοσλαβία και ξαναχάρασε τα σύνορα στην περιοχή με το αίμα των λαών της που ενίσχυσε το εθνικό μίσος και τις διαιρέσεις που δημιούργησε δύο άθλια προτεκτοράτα τη βοσνία και το κόσοβο που διατηρεί στη βοσνία παραπάνω από είκοσι χρόνια θέματα του νάτο του ευρωστρατού και της ιούλεξ. οι λαοί της βοσνίας κύριε πρόεδρε αυτό που έχουν ανάγκη δεν είναι η ένταξη στην ευρωπαϊκή ένωση αλλά η άμεση απομάκρυνση των στρατευμάτων κατοχή της ευρωπαϊκής ένωσης για να αποφασίσει ο λαός ελεύθερα την πορεία του. ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μια χώρα σαν τη Βοσνία Ερσεγοβίνη, πώς είναι δυνατόν να της δώσουμε το καθεστώς του υποψήφιου, της υποψήφιας χώρας προς ένταξη. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα διαφοράς, εγκληματικότητας. Είναι μια χώρα που έχει τεράστια τέτοια προβλήματα. Πριν από μερικέ εβδομάδες κάποιος από την ε, οικογένεια του Προέδρου συνελήφθη μαζί με 18 υπαλλήλους για διαφθορά. Ότι πήραν χρήματα από καταδικασμένους για να τους αθώσουν. Υπάρχει λοιπόν τεράστια διαφθορά, παθητική και ενεργητική, ναρκωτικά. Το οργανωμένο έγκλημα, με άλλα λόγια, είναι παρόν πάρα πολύ. Είναι μια τραγική κατάσταση αυτή με τη Σαρία επίσης, η οποία είναι παρόσα ο σύστημα στην Βοσνία Ζεγοβίνη. Νομίζω ότι φτάνει πια. Πρέπει να σταματήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με την διεύρυνση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πόσελτ. Κύριε Πρόεδρε, κανείς τις τελευταίες δεκαετίες δεν ασχολήθηκε με τη Βοσνία ζεγοβίνη δεν δεσμεύθηκε όπως η Ντόρι Πακ, η οποία πραγματικά έχει επισκεφθεί επανειλημμένο στην περιοχή αυτή και θα πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας αυτά που μας λέει σήμερα. Πιστεύω πραγματικά ότι αυτά που ακούμε για την αξιοπιστία, για τη διαφθορά, θα πρέπει να μας προβληματίσουν και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Θα ήταν σωστό να διαπιστώσουμε ότι ίσως έχουμε περιπλέξει λίγο την κατάσταση. Μια χώρα η οποία υπό την καθοδήγηση των Αμερικανών έχει λειτουργήσει τα τελευταία 20 χρόνια με ένα τελείως λανθασμένο τρόπο. Μήπως θα πρέπει αφού κουμπώσαμε λανθασμένο το πουκάμισό μας να το ξεκουμπώσουμε για να το κουμπώσουμε σωστά. Νομίζω μια τέτοια ε, ριζική αλλαγή δικαιολογείται. Και μια νέα ηγετική τάξη είναι απαραίτητη. Όλα αυτά θα πρέπει να τα σκεφτούμε γιατί έχουμε συνεισφέρει και έχουμε διαπιστώσει ότι η συνεισφορά μας οδήγησε σε αυτήν την κρίση. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι να επωφεληθούν οι πολίτες της Βοσνίας Ερσεγοβίνης από αυτές τις προσπάθειες. Χρειάζεται λοιπόν ανανέωση των δυνάμεων και των ελίτ αυτής της χώρας. Σας ευχαριστώ. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κ. Ζόλτσα για 1,5 λεπτό. Υπουργέ Επίτροπε, κανείς δεν περίμενε ότι η οδός ε, που θα ακολουθούσε η Βοσνία Ζεκοβίνη για να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν εύκολος ε, λόγω του, της ε, κληρονομιάς και της θεσμικής διάρθρωσης του κράτους. Φαίνεται ξεκάθαρα στο ψήφισμα της κυρίας Πάκο ότι υπολείπεται σοβαρό έργο, συνταγματική μεταρρύθμιση, παραδείγματος χάρη για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και να αποφύγουμε την πολιτική παράλυση τώρα και στο μέλλον. Χωρίς εύρυθμα λειτουργούς ε, ε εύρυθμα ε, λειτουργούς θεσμούς ε, δεν μπορούμε να εξυγχρονίσουμε τη χώρα και να με την απόφαση φύνση Ε, πέρα από την σωστή πολιτική εκπροσώπηση, το κράτος δικαίου και το δικαστικό σύστημα έχουμε και άλλες πολύ μεγάλες προκλήσεις ε, στη Βοσνία Ερσεγοβίνη, όμως αυτό δεν μπορεί να είναι μια πρόφαση για έλλειψη δράσης. Το αντίθετο, η πολιτική ελίτε θα πρέπει να επιταχύνει τις προσπάθειές της ε, για να προσεγγίσει η χώρα την Ευρωπαϊκή Ένωση προς όφελος του λαού της Βοσνίας Ερσεγοβίνης. Το Μοντενέ, το Μαυροβούνιο έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο και τώρα βλέπουμε ότι η Πριστίνα και το Βελιγράδι έχουν βελτιώσει τις σχέσεις τους. Εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει να υπολείπεται αυτό η Βοσνία Ζεγοβίνη. Το θέμα δεν είναι να θέλουμε να βοηθήσουμε. Το θέμα είναι οι τοπικοί ηθήνοντες να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ο Earl of Dartmouth, παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Βοσνία έχει μια φοβερή ανεργία, 43%. Είναι άλλη μια πάρα πολύ φτωχή ανατολική χώρα η οποία έχει μπει στο δρόμο ένταξης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άπαξ και ανοίξει η πόρτα στη Βοσνία, τότε θα υπάρξει τεράστια ροή ανθρώπων οι οποίοι θα πλημμυρίσουν μεταξύ άλλων το Ηνωμένο Βασίλειο που θα είναι και ο κύριος Μαγνήτης για αυτούς. Το Συνταγματικό Κόμμα στο Ηνωμένο Βασίλειο λέει ότι θέλει να μειώσει τη μετανίστευση. Όμως όπως γνωρίζουμε όλοι δεν είναι δυνατόν αυτό όσο παραμένουμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως χώρα. Και η αδυναμία αυτή θα γίνεται όλο και μεγαλύτερη όσο περισσότερες χώρες μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όσο οι άνθρωποι, οι πολίτε του έχουν δικαίωμα της ελεύθερης διακίνηση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα και να μπαίνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κανείς λοιπόν δεν μπορεί να στηρίξει την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Βοσνίας Ερζεγοβίνη, από όπου και αν προέρχεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πόστελ έχει ε, μπλε κάρτα προς τον κύριο Ρούτζεκ. Δέχεστε να απαντήσετε. Κύριε Πόσελτ, σας ακούμε. Ευχαριστώ. Ήθελα να πω στον κύριο Ρότσεκ, πριν από λίγες εβδομάδες η Κροατία πήγε στην τελική φάση της προσχώρησης ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για μια χώρα που έχει κάποιες ε, διασυνοριακές διαφορές εδαφικές με την Βοσνία Ζεγοβίνη. Η περιοχή της Μπάνια και άλλες σήμερα βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της αμφισβήτησης. Α, δύο μπλε κάρτες. Να απαντήσω σύντομα σε αυτήν την ερώτηση. Ναι, ναι, καταλαβαίνω και βλέπω δυνατότητες ε, πρέπει να υποστηρίξουμε αυτήν την προσπάθεια η Βοσνία Ζεγοβίνη και για τους πολίτες ε, αυτής της χώρας σίγουρα θα επιδεινωθεί η κατάσταση όταν μπει η Κροατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σίγουρα θα δυσκολέψει η κατάσταση για αυτούς που θέλουν να ταξιδέψουν στην Κροατία και φυσικά και όσον αφορά το εμπόριο θα υπάρξουν κάποια, κάποιες αλλαγές. Αλλά εμείς πρέπει να ενισχύσουμε αυτήν την διασυνοριακή ε, εμπορική συνεργασία. Τον κύριο Ντόρτμουθ, μπορώ να τον ρωτήσω κάτι. Μπορείτε να μας δώσετε ένα νούμερο. Γιατί εσείς παρουσιάσατε τον λαό της Βοσνίας Ερζεγοβίνης σαν ε, μια διεφθαρμένη χώρα η οποία έχει 62-63 εκατομμύρια. Μπορείτε να μας δώσετε ένα νούμερο να μας πείτε πόσοι από τη Βοσνία Ζεγοβίνη κατά τη γνώμη σας ζουν αυτή τη στιγμή στον Ηνωμένο Βασίλειο. Ότι θα κατακλείσουν το Ηνωμένο Βασίλειο που έχει 63 εκατομμύρια κατοίκους. Νομίζω ότι δεν καταλάβατε. Δεν λέω ότι τώρα είναι πολύ, αλλά ακριβώ αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί προς το παρόν ελέγχουμε την μετανάστευση από τη Βοσνία Τζεγοβίνη. Έτσι και γίνει η χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βοσνία Τζεγοβίνη, δεν θα μπορούμε πια να ελέγχουμε. Εσεί και οι συνάδελφοί σα το έχετε πει αυτό πολλέ φορέ. Και με στήριξη μάλιστα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα γίνεται αυτό. Κύριε, κύριε Ντάρτμουντ, έχουμε και άλλη μπλε κάρτα. Από την κυρία Κορνέλισεν. Δέχεστε. Παρακαλέστε το λόγο, κυρία μου. Κύριε Ντάρτμουν, στην παρέμβασή σας φάνηκε ότι αύριο θα γίνει μέλος η Βοσνία Ερζεγοβίνη. Δεν νομίζω να συμβεί αυτό. Υπάρχει μια διαδικασία για την προσχώρηση και χρειάζονται μεταρρυθμίσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δίκαιου, της οικονομικής συνεργασίας, ε, Τη ανταγωνιστικότητα ε, για την ένταξη στην ενιαία αγορά δεν το επιθυμείτε. Αυτό για τους πολίτες τη Βοσνίας Ερζεγοβίνη δεν θέλετε να, έχετε αυτό, να έχουν αυτό το όραμα των μεταρρυθμίσεων. Ε, αγαπάτε αλλήλους, αυτό ισχύει μόνο για τους Βρετανούς υπήκοου και για κανέναν άλλον. Απάντηση. Ε, είχα την εντύπωση ότι ήμουν σαφέστατος, ε, πέραν του δέοντος, ότι είμαστε κατά της προσχώρησης Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Πέραν αυτού αντιτασσόμεθα και στην ε, Μακεδονία και στην Σερβία και κυρίως την προσχώρηση της Τερκίερ, πέρα από την Αλβανία και το Μαυροβούνιο. Είμαστε κατά της προσχώρησης όλων αυτών των χωρών. Ε, αυτό είναι ένα και βασικό. Α, και εντάγει να σας πω και το εξής ότι αν ήταν για αύριο η προσχώρηση μπορείτε να πείτε ε, αργήσατε και δεν αντιταχθήκατε εγκαίρως. Ε, λοιπόν γι' αυτό εμείς αντιδρούμε εκ των προτέρων για να είναι εγκαίρως. Ε, ο επόμενο ε, ομιλητή είναι ο κύριος Μέλτζερ. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε με τη Βοσνία έχουμε μια κλασική περίπτωση ενός κεντρικού κράτους με πολύ δυνατές περιοχές. Το θέμα είναι ότι αυτό που απαιτείται για να υπάρξει διακυβέρνηση είναι περισσότερη συγκέντρωση εξουσίας. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την κατάσταση που συμβαίνει εκεί. Εδώ και χρόνια η Βρυξέλλες έχει πει έχουν πει ναι σε κάποια πράγματα τα οποία βλέπουμε δεν φέρνουν απολύτως κανένα αποτελέσματα. Τώρα όσον αφορά το θέμα των συνόρων, είναι ιερά αυτά τα σύνορα και δεν πρέπει να τα ε, αγγίξει κανείς. Καταλαβαίνετε όμως ότι η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τώρα δεν έχει αποφέρει τα αποτέλεσμα. Συνεχίζουν να υπάρχουν διακρίσεις, παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βλέπουμε ότι οι Σέρβοι που ζουν στη Βοσνία είναι θύματα πολλών τέτοιων παραβιάσεων. Αυτή λοιπόν η κεντρική εξουσία θα πρέπει να μπορέσει να προστατεύσει όλους και όχι μόνο τους μουσουλμάνους Βόσνιους. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος ομιλητής η κυρία Μπασέσκου. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Στηρίζω την ε, διεύρυνση προς Ανατολάς της Ευρώπης και προς τα Βαλκάνια, τα Δυτικά Βαλκάνια, τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως η Βοσνία Ριζεγοβίνη είναι η μόνη χώρα στην περιοχή όπου δεν υπήρξε επαρκής πρόοδος στην διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και ο κύριος λόγος είναι ότι δεν υπάρχει αρκετό όραμα όταν πρέπει να επιλέξει το δρόμο της η χώρα. Η διοίκηση της χώρας έχει σαν αποτέλεσμα οι αποφάσεις να καθυστερούν πάρα πολύ. Υπάρχουν αμφιβολίες για τις δυνατότητες λοιπόν που έχει η χώρα αυτή να λειτουργήσει ως πραγματική χώρα. Και οι πολιτικοί και οι πολίτες έχουν τις αμφιβολίες αυτές. Πάντως οι αποκλήσεις που υπάρχουν ανάμεσα στους πολιτικούς και τα συμφέροντα της χώρας είναι αυτό το οποίο εμποδίζει τελικά ε, το να προχωρήσει η χώρα και να φτάσει να γίνει μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είτε πρόκειται για τη διεύρυνση προς Ανατολασί, είτε πρόκειται για τη διεύρυνση προς τα Δυτικά ε, Βαλκάνια, δεν μπορεί να επιτευχθεί συνένεση. Το θέμα των μειονοτήτων επίσης είναι πολύ ανισχυτικό. Το Σύνταγμα επιτρέπει μόνο στους Βόσνιους Σερβοκροάτες να μπορούν να είναι υποψήφιοι στις προεδρικές εκλογές ή για το Κοινοβούλιο. Επίσης θέλω να πιστήσω την προσοχή σας και στον σκεπτικισμό που επικρατεί απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που θα διευρυθεί και στον πληθυσμό. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Φαγιόν έχει τώρα το λόγο. Η κυρία Φαγιόν για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εδώ πρέπει να πούμε πραγματικά ότι υπάρχει η πολιτική παραλυσία στην Βοσνία Ριζαγοβίνη. Οι υποσχέσει δεν έχουν τηρηθεί, οι μεταρρυθμίσεις δεν έχουν γίνει και οι επιπτώσεις είναι σαφείς σήμερα για όλους. Θα ήθελα επίσης να πω ότι η σημερινή κατάσταση μας δείχνει πώς έχει η κατάσταση επιτόπου δεν μπορούμε όμως με μια τόσο ριζοσπαστική πρόταση όπως αυτή του αποκλεισμού της βοσδίας Ερζεγοβίνης από το Συμβούλιο της Ευρώπης να λύσουμε τα προβλήματα. Υπάρχει πολιτική κρίση η οποία θα ακολουθήσει ουσιαστικά τις υπόλοιπες κρίσεις που μαστίζουν τη χώρα αυτή. Φοβάμαι πάρα πολύ ότι μια τέτοια πρόταση θα μας οδηγήσει προς την τελείως λανθασμένη κατεύθυνση και μπορούμε πραγματικά να αποτελέσουμε παράδειγμα για τις μεταρρυθμίσεις σε αυτή την περιοχή. Όσον αφορά τώρα την προσχώρηση της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό σίγουρα για τον άμεσο γείτονα της Κροατίας στην Βοσνία Ριζεγοβίνη, θα έχει κάποιες επιπτώσεις. Αυτές τις έχει ήδη περιγράψει η Ιρλανδική Προεδρία και πιστεύω ότι για τους πολίτες της Βοσνίας της Ζεγοβίνης παραδείγματο χάρη η μετακίνηση προς την Κροατία θα δυσκολέψει. Δεν μπορούμε όμως σήμερα εμείς να τιμωρήσουμε τους πολίτες της Βοσνίας της Ζεγοβίνης για τα σφάλματα των πολιτικών της πολιτικής ηγεσίας. Εδώ πραγματικά κινδυνεύουμε να τιμωρήσουμε τους πολίτες της Βοσνίας της Ζεγοβίνης με αυτά τα μέτρα. Κούκαν. Ευχαριστώ. Θα πω κάτι που δεν έχει πει κανένας μέχρι τώρα. Θέλω να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Φίλε και την Αντιπρόεδρο Άστον για την στήριξή τους στις μεταρρυθμίσεις στην Βοσνία. Βέβαια, είναι αλήθεια ότι οι συζητήσει που κάνουμε είναι όλο και πιο απογοητευτικέ. Είναι θλιβερό το γεγονό ότι οι ευρωπαϊκέ φιλοδοξίε τη χώρα αυτή και των πολιτών τη παραλύονται τόσο συχνά εξαιτία των ε, τοπικών πολιτικών και την ανικανότητά τους να καταλήξουν σε λύσεις όταν πρόκειται για τις βασικές αρχές λειτουργίας μιας χώρας. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν είναι να αναλάβει την ευθύνη για τις εξελίξεις στην Βοσνία, οι τοπικοί πολιτικοί θα πρέπει και εκείνη να αναλάβουν τις δικές τους ευθύνες για την τρέχουσα κατάσταση. Και εδώ μιλάω κυρίως για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πώς είναι δυνατόν τέσσερα χρόνια μετά την απόφαση του δικαστηρίου στην υπόθεση Φίντσι ακόμα να μην έχουμε δυνατότητα να αλλάξουμε το Σύνταγμα έτσι όπως πρέπει και να μπορούν όλοι οι πολίτες να είναι υποψήφοι για την τα νότατα αξιώματα της χώρας. Μα είναι προϋπόθεση για οποιαδήποτε χώρα θέλει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάω για τη φιλοδοξία της Βοσνίας Ερσεγοβίνης να ενταχθεί στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Η τελευταία έκθεση που έχουμε για την πρόοδο της χώρας μιλάει για περιορισμένη πρόοδο και για καθόλου πρόοδο. Μα η βασική προϋπόθεση για το μέλλον, για οποιαδήποτε πρόοδο της χώρας αυτής, είναι να μπορούν να ε, μιλήσουν με μία φωνή οι Βόσνοι, ενωμένοι. Δεν χρειάζονται μεταρρυθμίσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση, χρειάζονται μεταρρυθμίσεις για τον λαό της χώρας αυτή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει, αλλά την ευθύνη την έχουν εκείνοι στα δικά τους τα χέρια, οι ντόπιοι πολιτικοί δηλαδή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Έξι έχουν ε, ζητήσει να πάρουν το λόγο στη διαδικασία Catch the Eye. Θα πάρουν το λόγο και οι έξι, εφόσον τηρούν βέβαια το χρόνο ομιλία τους, που είναι ένα λεπτό. Ο πρώτο είναι ο κύριο Μπάνκινγκ. Ε, σας ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές. Η Βοσνία Ζεγοβίνη έχει περιέλθει σε εξαιρετικά δεινή κατάσταση διότι ε, είναι ευάλωτη όπως και άλλα ομόσπονδα κράτη. Οι τρεις εθνοτικές ομάδες ε, συνυπάρχουν σε αυτή τη χώρα και ήδη είναι δύσκολη όσο έχει η κατάσταση. Εγώ ε, ζούσα στον νότο της Ουγγαρίας και υπάρχουν ε, Κροάτες, ε, Σέρβοι, Γερμανοί και άλλες ομάδες που οι ειρηνικά και η πόλη του Πίτσε βρίσκεται στην ίδια κατάσταση. Η Ουγγαρία όμως ενεπλάκει και επεδίωξε να σταθεροποιηθεί η κατάσταση στην Βοσνία Ζεγοβίνη το ταχύτερο δυνατόν. Επιδίωξε την επιτάχυνση της διαδικασίας ε, της προσχώρησης ε, για να επιταχυνθούν και οι διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε λοιπόν να υιοθετήσουμε τώρα διαφορετική στάση, διότι πρόκειται για την νότια απειλή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Κροατία ε, μετά την προσχώρησή της θα διευκολύνει τη διαδικασία. Σας ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος, ο κ. Βαντερχότσεν. Ευχαριστώ πολύ. Πιστεύουμε ότι πρόκειται για μια κατάσταση πραγματικά τραγική. Με το τέλος του πολέμου δίνουμε πια όλο και λιγότερη προσοχή στις χώρες αυτές. Και είναι άδικο αυτό, δεδομένου ότι υπήρξαν τόσα θύματα. Η χώρα αυτή έχει σταματήσει. Κάθε ελπίδα να βγούμε... Δεν υπάρχει καμία διέξοδος από το αδιέξοδο. Αυτό όμως δεν πρέπει να μας οδηγήσει στο να τα παρατήσουμε. Σημαίνει αυτό πως ε, έχουμε καταλήψει κάθε ελπίδα από αυτές που γεννήθηκαν μετά τον πόλεμο. Η κατάσταση θα αλλάξει όταν δώσουμε περισσότερη προσοχή στην Βοσνία Ζηγοβίνη και ασκήσουμε την απαραίτητη πίεση για να βρεθούν λύσεις. Πάνω απ' όλα δεν επιτρέπεται να αφήσουμε τη χώρα μόνη της. Αλλιώς θα την αφήσουμε στους εξτρεμιστές. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Κάτσιν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριε Επίτροπε. Επ' ευκαιρία της ένταξης της ε, Κροατίας, το Συμβούλιο θα πρέπει να ενθαρρύνει την Βοσνία Ζεγοβίνη να διατηρήσει τις ρυθμίσεις συνοριακές που έχει μέχρι και μετά την 1η ε, Ιουλίου, καθώς ε, η Κροατία εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι στη ζώνη Σέγγεν. Πρέπει να δείξουμε αλληλεγγύη με τους Βόσνιους πολίτες και να βοηθήσουμε στην οικονομική ανάπτυξη και να ευνοήσουμε τις επαφές των ανθρώπων. Ταυτόχρονα πρέπει να διαφωνήσω με την τροπολογία 7 που ζητάει από το Συμβούλιο της Ευρώπης να αναστείλει την ε, ιδιότητα μέλους της Βοσνίας. Δεν πρέπει να απομονώσουμε περαιτέρω τη χώρα, αλλά να τη βοηθήσουμε δεν πρέπει να την ταυτίζουμε με τη Λευκορωσία, τη μόνη ευρωπαϊκή χώρα που δεν είναι μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης. Νομίζω αυτό παραπάει. Πρέπει τέτοιες τροπολογίες να συζητιούνται πρώτα στην Επιτροπή Εξωτερικών. Πρέπει να τίνουμε χείρα βοηθείας στους Βόσνιους πολίτες και θα πρέπει η χώρα να πάρει τη μοίρα της στα χέρια της. Ευχαριστώ. Σας ε, ευχαριστώ. Ο κύριος Πάσκα για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Βοσνία Ριζεγοβίνη είναι η χώρα με την πιο πολύπλοκη πολιτική δομή στα Βαλκάνια. Είναι διχασμένη εθνικά και θρησκευτικά και δεν μπορούν να λειτουργήσουν άρα κρατικές δομές. Οι μνήμες του πολέμου είναι πρόσφατες και άρα υπάρχει μεγάλος βαθμός δυσπιστίας μεταξύ των ηγετών των διαφόρων κοινοτήτων της ε, χώρας. Ε, η Κροατία και η Σερβία βεβαίως με το παράδειγμα τους δείχνουν πως μια λογική και ειρηνική επίλυση των προβλημάτων χωρίς προκαταλήψεις μπορεί να αποτελέσει τον τρόπο προόδου αυτής της χώρας. Οπότε πρέπει να συνεχιστεί η διαδικασία ολοκλήρωσης στα Βαλκάνια και να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του πληθυσμού της χώρας αυτής. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση παρά το ότι είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Σας ευχαριστώ. κύριος Μπρόνς. Εγώ συγχαίρω τη Βοσνία Ερζεγοβίνη που δεν έχει κάνει πρόοδο προς την ε, επίτευξη των πολιτικών κριτηρίων. Όσο πιο πολύ αντισέκεται μια χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο το καλύτερο. Ειδικά δε η αντίστασή της ε, στην ε, νεοφιλελεύθερη οικονομία και αυτό σε αντιδιαστολή με την οικονομία των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Βεβαίως ήμουν ε, έτοιμος να τους ε, συγχαρώ όταν μίλησαν για ελευθερία διακίνησης, αλλά ενώσαν ελευθερία διακίνησης μέσα στην ίδια τους τη χώρα. Αν είναι κανείς Κροάτης θα το ξανασκεφτεί να περάσει από τη Ρεπούμπλικα Σέρβσκα. Οπότε ο πληθυσμό είναι χωρισμένος στα τρία, η πολιτική συνεργασία δεν υφίσταται. Θέμε πραγματικά μια τέτοια διχασμένη χώρα να ενταχθεί στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως Ξέρουμε πω μια χώρα διχασμένη ε, είναι ακυβέρνητη, Όπω φαντάζομαι συμπεραίνουν αυτή τη στιγμή και οι Σουηδοί στη Στοκχόλμη. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω για την συζήτηση αυτή. Είναι μια συζήτηση η οποία δείχνει ότι η κατάσταση στη Βοσνία Ερσεγοβίνη δεν είναι ικανοποιητική για κανένα μας. Το θέμα όμως που τίθεται και είναι θεμελιώδες είναι το εξή. Τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι η χώρα δεν πρέπει να έχει την προοπτική να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τη γνώμη μου πρέπει να έχει μια τέτοια προοπτική, διότι αλλιώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χάσει ένα σημαντικό μέσο επιρροής τη κατάστασης στη χώρα. Όταν συζητάμε για τη χώρα αυτή πρέπει να έχουμε υπόψη μας και το ιστορικό πλαίσιο και το εθνοτικό πλαίσιο. Νομίζω ότι είναι προτιμότερο να συνεχίσει η προσπάθεια της χώρας να προσαρμοστεί με όλες τις προδιαγραφές και όχι να την αφήσουμε στη μοίρα της. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Τώρα. Έχουμε φτάσει στο τέλος της συζήτησης αυτής. Το λόγο έχει ο Επίτροπος Φίλε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, Καμιά φορά μετανιώνω όταν αποκλίνω από το κείμενο που μου έχουν προετοιμάσει. Ελπίζω να μην το μετανιώσω και σήμερα. Ο κύριος βουλευτής που ανέφερε το ζήτημα της ελεύθερης διακίνησης ε, αψιάζει, οπότε δεν θα αναφέρθω ε, ονομαστικά σε αυτόν. Συνήθως, βεβαίως, καλό είναι να αποφεύγουμε τις προβλέψεις και ειδικά όσον αφορά την διαδικασία της διεύρυνσης. Θα γίνει μια εξαίρεση σήμερα όμως και ελπίζω οι συνάδελφοι να με συγχωρήσουν. Η Βοσνία δεν έχει ακόμα κάνει αίτηση για να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν λοιπόν είναι κατάλληλες οι συνθήκες, προβλέπω πως σε μερικούς μήνες θα ε, υποβάλει αίτηση, πρέπει να την εξετάσει το Συμβούλιο, θα έχουμε μία συμφωνία σύνδεσης ε, και μετά, αν όλα πάνε καλά, μπορεί να προτείνουμε την έναρξη διαπραγματεύσεων, μπορεί να έχουμε κάποιες διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις, θα υπάρξει ένας έλεγχος για ένα έτος, πέντε έτη διαπραγματεύσεων, δύο έτη διαδικασία κύρωσης, οπότε να σας υπενθυμίσω πως τα κράτη-μέλη έχουν 7 χρόνια μπροστά τους για να προστατεύσουν την εσωτερική τους αγορά ε, απέναντι στην ελεύθερη διακίνηση εργαζομένων. Αν όλα πάνε καλά. Μιλάμε για 17 χρόνια από σήμερα, έτσι. Ε, χρειάζεται όραμα για να προβλέψει κανείς το τι θα γίνει σε 17 χρόνια από σήμερα. Και να σου πω και δεν το βλέπω κιόλας με βάση την εμπειρία που είχαμε. Ε, είναι η χώρα την οποία γνωρίζω καλύτερα μετά το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου ήμουν ε, πρεσβευτής. Τρία πράγματα τώρα έχουμε. Ε, ευθύνη απέναντι στην ε, Βοσνία. Το Dayton το 1995 τους επιβάλαμε μια συμφωνία. Έχουμε μια δέσμευση αναλάβει. Η συμφωνία αυτή του Dayton ήταν το καλύτερο πλαίσιο για να μπορέσει η Βοσνία να έχει φτάσει λοιπόν η στιγμή να σκεφτούμε ένα άλλο πλαίσιο τώρα για να μετασχηματιστεί η Βοσνία Ριζεγοβίνη. Η διεύρυνση είναι το πιο ισχυρό μέσο που έχουμε. Δεν είναι Dayton, είναι διεύρυνση. Μέσω της διεύρυνσης θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε κάποια από αυτά τα ζητήματα για τα οποία παραπονιέστε και εμείς παραπονιόμαστε. Χρειάζεται να του βοηθήσουμε να περάσουν αυτή τη γέφυρα, να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η γέφυρα αυτή Η απόφαση αυτή ήταν λοιπόν ε, Σέντι Βίντσι. Αφορούσε στην ε, διαδικασία στη χώρα αυτή. Τι κάνουμε λοιπόν. Θα βρεθεί η Βοσνία ζεγοβινη στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δείχνει η Πριστίνα και Βελιγράδη τον δρόμο. Και δείχνει πόσο σημαντική είναι η ευρωπαϊκή προοπτική και τι δυνατότητες υπάρχουν. και τι μπορεί να επιτύχει η διεύρυνση. Οπότε πρέπει να βοηθήσουμε την ε, Βοσνία που παραμένει η μόνη χώρα η οποία περιμένει μόνη της στο κρύο στο, στο πλαίσιο του Dayton ενώ όλες οι υπόλοιπες χώρες προχωρούν προς το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα το τρίτο στοιχείο. Καμιά φορά αναφερόμαστε στην απόφαση Σέιντιτς Φίντσι ως το μοναδικό εμπόδιο στην αίτηση ένταξης. Δεν ισχύει αυτό. Η Σέιντιτς Φίντσι είναι ο λόγος για τον οποίο δεν έχουμε την εφαρμογή της Συμφωνίας Σύνδεσης. Γιατί την ε, επόμενη μέρα εάν ε, τεθεί δηλαδή σε ισχύ αυτή η συμφωνία θα πρέπει να ξεκινήσουμε διαδικασίες επί παραβάση. Η Βοσνία Ερσεκοβίνη δεν συμμορφώνεται με τις διεθνείς της δεσμεύσεις. Και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Και έρχομαι εδώ πέρα άρα στο ψήφισμά σας και στις σχετικές ε, τροπολογίες. Τώρα δεν μπαίνω συζήτηση για το εάν μία ε, η υψή πρόταση είναι η σωστή. Αλλά συμφωνώ πως έχει φτάσει η ώρα για να χτυπήσει ένα καμπανάκι. Ναι, έχει φτάσει αυτή τη στιγμή. Και ενώ άκουσα πολλούς από εσάς να αναφέρεστε σε αυτή την ε, τροπολογία και να λέτε πως δεν θα την στήριξετε. Ε, δεν άκουσα κάποια εναλλακτική πρόταση. Δεν άκουσα κάτι. Δεν άκουσα μία πρόταση για το πώς θα επιτρέψουμε στη Βοσνία Ζεγοβίνη να ανταποκριθεί στις διεθνείς της ε, δεσμεύσεις. θα, έχουμε, θα έχουν βουλευτικές εκλογές σε λίγους μήνες. Του χρόνου δηλαδή. What if we have uh, another... Τι θα κάνουμε τότε, τι θα γίνει αν έχουμε και άλλες βουλευτικές εκλογές στη Βοσνία Ζεκοβίνη χωρίς να ε, υπάρξει συμμόρφωση με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Θα περιμένουμε τότε να χτυπήσει καμπανάκι. Ε, τώρα είναι η στιγμή όχι να απειλήσουμε αλλά να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα. Πρέπει να δουν τι θα κάνουν με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, να ευθυγραμμίσουν το Σύνταγμά τους με την απόφαση αυτή Αλλιώς, όχι μόνο δεν θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση ένταξη, αλλά θα έχουν παραβιάσει και τις ε, διεθνείς τους υποχρεώσεις. Και αυτό έχει συνέπειες. Uh, Μεταξύ και των οποίων βεβαίως και η προσωρινή εφαρμογή της ε, Συμφωνίας ε, Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. Και το δεύτερο σαφές μήνυμα είναι πως είμαστε εδώ να σας βοηθήσουμε γιατί είμαστε εταίροι σας. Έχουμε δείξει πόσο σοβαροί είμαστε, θέλουμε να σας βοηθήσουμε να περάσετε αυτή τη γέφυρα. Εντάξει. Αν δεν κάνουμε εμείς αρκετά, θα διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας. Αλλά χρειάζεται και αυτό το κοινό όραμα από εσάς. Γιατί σε τελική ανάλυση εσείς πρέπει να ανταποκριθείτε στις προσδοκίες των πολιτών σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Από πλευράς του Συμβουλίου, κυρία Κρέιτον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Φυσικά, η συζήτηση ήταν ε, λυπηρή, γιατί υπάρχει μια διάχυτη αίσθηση απογοήτευσης. Όμως νομίζω ότι ήταν και ιδιαίτερα επικοδομητική και βοηθητική συζήτηση και για την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Να επαναλάβω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απόλυτα και απαράβατα αφοσιωμένη στην ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Ας το δούμε από λίγο παλιότερα. Να θυμηθούμε ότι οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα έχει δικαίωμα να γίνει μέλος της Ένωσης εφόσον πληρεί τα κριτήρια. Δεν είναι λοιπόν θέμα τα, μέλλον, τα, συγγνώμη, τα παρόντα να αποφασίσουν εάν και κατά πόσον κάποια άλλα κράτη μέλη της Ένωσης θα ενταχθούν. Είμαστε όλοι δεσμευμένοι. Είμαστε όλοι δεσμευμένοι και ιδιαίτερα δεσμευμένοι υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Όχι μόνο με βάση τη διακήρυξη της Θεσσαλονίκης για την οποία θα γίνει μια ειδική διάσκεψη της Προεδρίας την Παρασκευή στο Δουβλίνο όπου θα συμμετάσχει και η Επιτροπή. Αλλά όπως είπε και ο Επίτροπο Φίλε, επίσης η δέσμευσή μας δεν είναι μόνο δέσμευση, είναι και ευθύνη γιατί είμαστε εταίροι με βάση τη συμφωνία του Ντέιτον. Πρέπει να το έχουμε αυτό πάντα στο νου μας. Ως ε, ε, ε, παράγοντες στη διεθνή σκηνή έχουμε ευθύνη προς όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και ιδιαίτερα έναντι μιας χώρας όπως η Βοσνία Ζεγοβίνη όπου υπάρχουν τόσες διαιρέσεις και όπου ακόμη να αντιμετωπίσουν τόσες προκλήσεις, τόσα εμπόδια για να μπορέσει ο λαός της χώρας αυτής να ζει εν αρμονία, να επανενωθεί στα πλαίσια της ευρωπαϊκής οικογένειας. Όπως είπα η Ένωση θα συνεχίσει να βοηθάει τη χώρα θα ενισχύσουμε την παρουσία μας επιτόπου, σαφής δέσμευση εκπεφρασμένη, αλλά συμφωνώ με τα πολλά μέλη συμπεριλαμβανομένης της κυρίας Πακ και της κυρίας Μπόσκουρ, του κυρίου Κούκαν και πολλών άλλων που είπαν ότι η ευθύνη για να υπάρξει πρόοδος είναι θέμα των ηγετών και των θεσμών της. Αυτό πάντα ισχύει για όλες τις χώρες. Η Ένωση μπορεί να βοηθήσει, επικοδομητικά, να συμβάλλει, αλλά δεν μπορούμε να υποκαταστήσουμε τις ενέργειες που απαιτείται να αναλυφθούν από την πολιτική ηγεσία της ε, χώρας. Ε, είναι ζωτικές οι μεταρρυθμίσεις. Αντίθετα από ό,τι ε, είπε ένας παρεμβαίνων, οι μεταρρυθμίσεις αυτές βασίζονται στο δικό μας σύστημα αξιών. Οι αξίες αυτές είναι ο σεβασμός της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των μειονοτήτων, το κράτος δικαίου. Αυτές είναι αξίες στις οποίες βασίζεται η ίδια η Ένωση. Σωστό λοιπόν και πρέπει να εργαστούμε μαζί τους, να τους ενθαρρύνουμε, τους συνευρωπαίους μας ακόμη και αν ανήκουν στην Ένωση, να προσβλέπουν στην εφαρμογή αυτών των αξιών στο εσωτερικό της χώρας τους για το καλό των πολιτών τους. Και δεν απολογούμε γι' αυτό. Δεν απολογούμε σε κανέναν. Που επιμένω ότι πρέπει αυτοί οι κοινοί μας στόχοι να επιδιωχθούν και να επιτευχθούν. Είναι λοιπόν αναγκαίες αυτές οι μεταρρυθμίσεις κλειδιά, όχι επειδή εμείς καλούμε για αυτές, γιατί είναι φανερό ότι είναι προς το συμφέρον της χώρας και των πολιτών της. Σωστά υπόθηκε ότι όλα αυτά δεν θα γίνουν σε μια μέρα. Δεν χρειάζεται να φοβόμαστε τίποτα. Δέκα χρόνια έχουν περάσει από τότε που η Κροατία ξεκίνησε το ταξίδι της προς την ένταξη στην Ένωση και με χαρά διαπιστώνουμε όλοι ότι την 1η Ιουλίου αυτό το ταξίδι θα έχει λήξει. Οι άλλες χώρες της περιοχής σημειώνουν πρόοδο. Ιδιαίτερα όπως είπαμε πριν από δύο εβδομάδες στην περίπτωση της Σερβίας και του Κωσυφοπεδίου και η εργασία της ε, κυρίας Άστον, του κυρίου Φιούλε και άλλων οπωσδήποτε έχει βοηθήσει. Του συγχαίρουμε για την αφοσίωση και αιμονή με την οποία κατέληξαν σε αυτή τη συμφωνία, αλλά έχουμε ακόμη πολύ δρόμο να διανύσουμε. Για όλες τις άλλες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Αλλά είμαστε αποφασισμένοι να σημειωθεί πρόοδος ούτω ώστε να γίνει πραγματικότητα η δέσμευση που κάνουμε προς αυτού τους συνευρωπαίους μας. Είπαμε ότι θα γίνει αυτή η διάσκεψη στο Δουβλίνο για την διακήρυξη Θεσσαλονίκη καλή ευκαιρία όλοι εμείς οι Ευρωπαίοι να συζητήσουμε. Όπως και χθες κάναμε μια συζήτηση εδώ στην Ολομέλεια. Αναφερθήκαμε στο γεγονός ότι πάντα μπορούμε να επιδιώκουμε και να μας αρέσουν οι ιδανικές ουτοπικές καταστάσεις. Αλλά στην περίπτωση της διεύρυνσης με τα Δυτικά Βαλκάνια πρέπει να θυμηθούμε το σημείο αφετηρίας να θυμηθούμε την αιματοχυσία, τους πολέμους, τις τραγωδίες που έγιναν εδώ μπροστά στο κατόφλι μας. Πολύ πρόσφατα. Και πόση πρόοδος να αναλογιστούμε έχει σημειωθεί έκτοτε στην περιοχή. Αυτή η πρόοδος είτε αφορά την Κροατία, είτε αφορά το Μαυροβούνιο, τις άλλες ε, χώρες που αργά αλλά σταθερά βαδίζουν την οδό προς την ένταξη στην Ένωση. Όλες αυτές οι χώρες είμαι πεπισμένοι ότι θα σημειώσουν παρόμοια πρόοδο οι άνθρωποι και στη Βοσνία. Βεβαίω είμαστε απογοητευμένοι. Θέλουμε να υπάρξει περισσότερη προσπάθεια από την ηγεσία, αλλά σίγουρα θα υπάρξει πρόοδο. Ευχαριστώ το Κοινοβούλιο για την ε, αφοσίωση που έχει επιδείξει για το θέμα αυτό. Η εργασία των εισηγητών πολλέ φορέ περνάει απαρατήρητη, αλλά είναι αυτοί οι οποίοι έρχονται σε επαφή με την κοινωνία των πολιτών, με τους πολίτες εκεί, με τα πολιτικά κόμματα με τις κυβερνητικές υπηρεσίες. Η εργασία σας έχει τεράστια αξία και συνεχώς ενισχύει το μήνυμα ότι υπάρχει ανάγκη μεταρρυθμίσεων και ότι θα υπάρξουν πολλές αμοιβέ αν σημειωθούν αυτές οι πρόοδοι για τους πολίτες, για τη χώρα. Η πρόταση της κυρίας Πακ τροπολογίας για να ανασταλεί η συμμετοχή ε, ε, στο δικαστήριο. Εγώ δεν έχω θέση το Συμβούλιο γι' αυτό, μπορώ προσωπικά μόνο να μιλήσω. Καταλαβαίνω βέβαια γιατί κάνετε αυτή την πρόταση. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει ανάγκη να υπάρξουν επιπτώσει για τι ενεργέ του. Αλλά από την άλλη μεριά το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πρέπει να είναι το σημείο προσφυγή για του πολίτε για να μπορούν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά του. Οπότε ανησυχώ ότι ίσω να έχει τα αντίθετα αποτελέσματα αυτή η πρόταση. Αλλά ε, να το συζητήσουμε περαιτέρω με το Κοινοβούλιο το θέμα αυτό. Ευχαριστώ και πάλι το Κοινοβούλιο. Ας θυμηθούμε όλοι πόσο σημαντικό είναι όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης να συνεργάζονται ούτω ώστε επικοδομητικά να βοηθήσουμε. Σε αυτή τη φάση η επίλυση, ή συγγνώμη, η λύση που προτείνεται και προτάθηκε και στο παρελθόν με τη συμφωνία του Ντέιτον προς τη χώρα αυτή και η δέσμευση που αναλάβαμε, η προοπτική που τους προσφέραμε για ένταξη, δεν λειτουργεί σε αυτή τη φάση. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Πρέπει λοιπόν να αφουγκραστούμε και τις προτάσεις που έκαναν οι Ρούτσεκ Πόσελτ και άλλοι για την ε, ουσιώδη ανάγκη συνταγματικής μεταρρύθμισης. Το ανέφερε και η Κομισιόν. Πρέπει να βαδίσουμε και προς αυτή την κατεύθυνση. Χρειαζόμαστε μια νέα προσέγγιση για τη χώρα αυτή. Υπάρχει συνένεση νομίζω μεταξύ μας εδώ σε αυτή την αίθουσα. Πρέπει να βρούμε νέα προοπτική που να σέβεται όλες τις κοινότητες, να σέβεται όλα τα άτομα που προέρχονται από, διαφορετική, από διαφορετικό σημείο κίνηση. Πρέπει να γίνει περισσότερη εργασία από την Επιτροπή, το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και προσβλέπω σε αυτή τη συνεργασία με όλου σα για να επιτύχουμε αυτό το στόχο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Έχει υποβληθεί πρόταση ψηφίσματος ε, για να καταλήξει η συζήτηση αυτή και γι' αυτό λίγη τώρα